το επόμενο θέμα στην ημερήσια διαταξή αμέσως ε, έχει γυρίσει συνήθεια στην υποεπιτροπή μας ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο ε, της Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Επιτροπής είναι πάντα ένας διακεκριμένος αρχηγός από ε, τις ένοπλες δυνάμεις ε, κάποιου κράτους μέλους και με ιδιαίτερη χαρά και τιμή καλωσορίζω τον στρατηγό Κλάουντιο Γκρατσιάνο, ο οποίος υπηρετεί σε αυτή τη σημαντική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική Επιτροπή στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο, τα καθήκοντα, τις προκλήσεις και προσπαθούμε να παραμένουμε ενήμεροι. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Στρατηγέ, χωρίς να μακρηγορώ περαιτέρω, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Έχετε λάβει όλα τα μέλη την αντίστοιχη τεκμηρίωση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά και η ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, στρατηγέ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κυρία Φωτίγκα. Αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα είναι τιμή η ευκαιρία που έχω να μιλώ ενώπιον σα, στου εκλεγμένου εκπροσώπου των πολιτών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σας ευγνωμονώ πολύ για την ευκαιρία που έχω να σα ενημερώσω για τη συμβολή τη Στρατιωτική μα επιτροπή στην Γενική ε, ΕΠΑ, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνα. Θέλω να εξαρώ το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η υποεπιτροπή σα. Είμαι εδώ με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης και δρώ ως εκπρόσωπος των αρχηγών επιτελείων και των 28 ε, κρατών μελών. Ταυτόχρονα είμαι και στρατιωτικός ε, σύμβουλος της ΥΠΑ της εκπροσώπους η Επιτροπή μας ε, στα πλαίσια αυτής της αποστολής ήταν και παραμένει προσιλωμένη ε, στην ε, χάραξη της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Συμμετέχουμε και στην χάραξη αλλά και στην εκτέλεση της συνολικής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένες συστάσεις και συμβουλές σε θέματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος για να βεβαιωθούμε ότι ε, ακούγεται η φωνή των τελικών χρηστών και των ικανοτήτων τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έχουμε στρατιωτική πραγματογνωμοσύνη ευρύτατη από τα κράτη-μέλη που μέσω της Επιτροπής μας ε, γίνεται ε, παροχή γερών και στιβαρών στρατιωτικών συμβουλών σε όλες τις φάσεις χάραξης και εκτέλεσης της ΕΠΑ. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις ε, που διεξάγονται χάρη στη συνεισφορά και την υποστήριξη των κρατών μελών και τρίτων χωρών σε κάποιες από τις πιο περίπλοκες και επικίνδυνες περιοχές του κόσμου είναι η βασική δραστηριότητα ε, της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής. Αυτό τον καιρό πολλές ένοπλες δυνάμεις από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στην άμεση γειτονία μας όπως είναι στα Βαλκάνια ή και μακριο, ε, μακρύτερα Σομαλία, Κεντρική Αφρική, Μαλή ε, όπως και στη Μεσόγειο, ε, στον κόλπο του Άντεν και αλλού. Ποιος είναι ο βασικός στόχος φυσικά η εστίαση είναι στην Αφρική θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργάζεται, γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να παράσχει ευημερία και ασφάλεια. Είναι πολλές οι απειλές και πολυδιάστατες. Θα ήθελα σύντομα να σας παρουσιάσω και να διευκρινίσω ε, τη δική μου ε, άποψη και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το πώς συνδέονται όλα αυτά και πώς επηρεάζουν απολύτως την αντίληψη που έχουμε. Υπάρχει και μια διαφάνεια που μπορεί να μας βοηθήσει. Ε, στα πλαίσια αυτά ε, ε, έχουμε μια τριγωνική σχέση που είναι μεταβλητή ε, ε, τρομοκρατία, μετανάστευση, αστάθεια. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις ασφαλείας, ε, στοχεύοντας συστηματικά τις τρεις αυτές μεταβλητές. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ε, τρομοκρατίας και μετανάστευσης. Ε, φυσικά οι μετανάστες δεν είναι σε καμία περίπτωση εγκληματίες, αλλά μπορούμε να περιορίσουμε τις συνέπειες της μετανάστευσης υποστηρίζοντας τις χώρες προέλευσης με μέτρα οικοδόμησης ικανοτήτων ή με μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Είναι ένα νέο είδος βοήθειας που παρέχουμε στην καταπολέμηση της νομοκρατίας ε, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Και είναι σαφές παράδειγμα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τις χώρες εταίρους για να δημιουργήσουν ικανότητες και να διαχειρίζονται τις κρίσεις τους μόνοι τους. Στη στρατιωτική πλευρά έχουμε τρεις εκτελεστικές και τρεις μη εκτελεστικές αποστολές. Η παλαιότερη εκτελεστική είναι η Αλτία, Αλθέα, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας γενικότερα στην περιοχή. Σε συνεργασία με, στα πλαίσια του Βερολίνου ΣΥΝ, που χρησιμοποιούμε κοινέ δομές σε στρατιωτικό επίπεδο και στρατηγικό επίπεδο. Ε, συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ ε, στα πλαίσια της ε, διατρατικής κοινότητας. Άλλη επιχείρηση, Αταλάντα, στον κόλπο του Άντεν, στον Ινδικό ωκεανό. Πολύ επιτυχή στη δεκαετία της ύπαρξής της για τις θαλάσσιες μεταφορές και άλλα σκάφη που είναι βάλωτα στην πειρατεία. Εκτός από την Αταλ... Ε, ε, η Αταλάντα είναι και σημαντική πλατφόρμα για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, όπως η Νότια Κορέα, που συμμετέχει συχνά και τακτικά με μια φρεγάτα ε, και συντονίζουμε δράσεις με την Κίνα, τις Ηνωμένε Πολιτείε και άλλες χώρες. Παραμένουν ανοιχτές αυτές οι δυνατότητες. αυτή τη στιγμή εδρεύει η Αταλάντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά τέλη Μαρτίου, λόγω και του Brexit, θα μετατεθεί η έδρα της στην ε, Ισπανία και κάποια στελέχη σταθμεύουν στη Βρέστη της Γαλλίας. Υπάρχει επιχείρηση Σοφία ε, στη Μεσόγειο για την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων ε, και των λαθρεμπόρων στη Μεσόγειο και σε συνεργασία με τη Λιβική Ακτοφυλακή ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις παράνομες δραστηριότητε ε, στα λιβικά χωρικά ύδατα ή στην επικράτεια της χώρας. Επίσης, ε, η Σοφία ασχολείται με την επιβολή εμπάργου στη εμπόριο όπλων. Και το, το τόνισαν πρόσφατα αυτό και οι Υπουργοί Αμήνης, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η Σοφία. Στο Μαλή, ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και Σομαλία είναι μη εκτελεστικού χαρακτήρα αποστολέ, είναι εκπαιδευτικέ για τι ένοπλε δυνάμει και συμβουλευτικέ προ τη στρατιωτική ηγεσία των χωρών. Ε, εξακολουθούμε να έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις και συνεργασία και είναι σημαντικό να αξιολογούμε το αποτέλεσμα εάν συνεισφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, στην συνολική εφαρμογή της παγκόσμιας Καθολική στρατηγικής. Έχουμε θετικά αποτελέσματα παρόλο που ήταν πολύ δυσμενείς οι συνθήκες, σε περίπλοκες και συχνά επικίνδυνες όπως σας είπα καταστάσεις, αλλά και παρά την πολύ περιορισμένη εντολή που έχουμε ε, σε σχέση με άλλες αποστολές ε, των Ηνωμένων Πολιτειών ή ε, των Ηνωμένων Εθνών που έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. η MPCC ήταν πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ο στρατιωτικός σχεδιασμός ε, και δυνατότητα διεξαγωγής ε, των αποστολών αυτών. Αυτό είναι ένα συντονισμό που γίνεται στι Βρυξέλλε κεντρικά έτσι ώστε να μπορούν ε, όσοι δρούν επί τόπου να αφιερωθούν στην αποστολή του. Συνεργαζόμαστε με τα Ηνωμένα Έθνη και την Αφρικανική Ένωση Ε, αλλά ο συντονισμός ε, δεν μπορεί να γίνει επιτόπου γιατί είναι πολύ λίγο το προσωπικό εκεί. στόχο μας είναι να διευρυνθεί η παρουσία εκεί για να έχουμε και μια μικρή εκτελεστική επιχείρηση ε, με μια μονάδα κοινού συντονισμού. Αυτή η κοινή προσέγγιση είναι κάτι που διαπιστώνουμε και στη συλλογή πληροφοριών, όπου χρησιμοποιούμε ε, πολιτικές και στρατιωτικές πηγές για να ενημερωνόμαστε και να γνωρίζουμε την κατάσταση. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε και νομίζω θα το συζητήσουμε ότι το MPC ε, δεν έρχεται σε αντίφαση με τις δομές διοίκησης ε, του ΝΑΤΟ και την ιεραρχία, ούτε αντικαθιστά τις δυνάμεις των εθνικών ενόπλων δυνάμεων. Εκτός από τις έξι αυτές αποστολές, έχουμε κάνει ε, πρόοδο ε, με συνένωση δυνάμεων, πόρων, οικονομικών και άλλων. Από την προσωπική μου εμπειρία μπορώ να σας πω, ως αρχηγός μιας πολυεθνούς ε, δύναμης από τάγμα μέχρι ε, ταξιαρχία στο Αφγανιστάν. Ε, ε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι αντιμετωπίζει ένας αρχηγός επιτόπου. Ε, επειδή δεν έχουμε οικονομικούς πόρους, ε, υπάρχει πρόβλημα διότι Υπάρχουν κανόνες και μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων που περιορίζουν και το, τη δράση μας και το αποτέλεσμα της. Παρά τα μεγάλα επιτεύγματα ε, που ε, κάνουν ε, οι αρχηγοί των αποστολών εκεί υπάρχουν αδυναμίες γιατί δεν μπορούμε να τους στείλουμε υποδομές και υλικό στις ένοπλες δυνάμεις τις οποίες εκπαιδεύουμε. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποια λύση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για την Ειρήνη. Και από την άλλη, αντιμετωπίζουμε και το εξής πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη δεν μας στέλνουν αρκετό προσωπικό και υλικό για να εκτελούμε τις αποστολές που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο 28. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. UTM Σομαλία. Λείπει 30% του απαιτούμενου προσωπικού και ε, προσεχώς θα φτάσουμε σε σημείο να μην μπορούμε να ε, εκτελούμε όλες τις αποστολές που έχουμε από ε, την εντολή μας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία οι εκπαιδευτές πηγαίνουν στο Μποάρ που είναι λίγο πιο μακριά από την ε, πρωτεύουσα αλλά δεν μπορούν να μετακινηθούν εκεί οι ένοπλες δυνάμεις αυτές και δεν υπάρχει και ιατρική υποστήριξη. Σε άλλες περιοχές έχουμε διπλό περιορισμό. Πρώτον, να πεμπλακούν οι διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεύτερον να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να δείξουν περισσότερη αλληλεγγύη και να δεσμεύσουν περισσότερους πόρους και ανθρώπινους και υλικούς. Θα ήθελα να τονίσω ότι ε, Ομόφωνα συμφώνησαν τα 28 κράτη-μέρη για τις αποστολές ΕΠΑ. Χρειάζεται μάλλον περισσότερη συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές φιλοδοξίες και τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται ε, να ε, εκτελεστούν αυτές οι αποστολές επιτόπου. Άλλη παρατήρηση. Τεχνικής φύσεως αυτή μάλλον. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της συχνά δραστηριοποιούνται παράλληλα ε, στην ίδια χώρα. Το Μαλί, α πούμε, είναι ένα καλό παράδειγμα. Έχουμε τη Μινούσμα από τα Ηνωμένα Έθνη, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιχείρηση Μπαρκάν ε, της Γαλλίας. Και τώρα έχουμε και τη νέα ομάδα των πέντε χωρών του Σαχέλ, το G5. Αυτό είναι ένα το παράδειγμα. Θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο σε στρατηγικό επίπεδο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιες συνθήκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να αποδίδει καλύτερα αποστολή μας. Πριν φύγω από τις αποστολές και τις επιχειρήσεις, θέλω να σας πω ότι έχουμε μια και άλλες αποστολές της CSDP στην ΕΠΑΑ και έχουμε και μια φιλοδοξία τώρα, διαφορετική συνεργασία πολιτικών στρατιωτικών δυνάμεων. Καλύτερη συνεργασία, κα, καλύτερο συντονισμός μεταξύ των δύο στοιχείων που είναι διακριτά μεταξύ τους αλλά συμπληρωματικά για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσεγγίζει εξωτερικές κρίσεις η μια πολιτική αποστολή ε, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της διάφορα στοιχεία σε ένα διεθνές περιβάλλον. Ο κάθε διεθνής οργανισμός έχει διαφορετικούς κανόνες διαχείρισης. Ας πούμε, τα Ηνωμένα Έθνη βάζουν υπό την ίδια διοίκηση ε, πολιτική και στρατιωτική αποστολή. Στο ΝΑΤΟ κυριαρχεί η στρατιωτική δομή, όπου ε, όλες οι μονάδες είναι από τη στρατιωτική ηγεσία και ιεραρχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο ε, έχει παράλληλες δομές στρατιωτικές και πολιτικές. Ε, ε, επειδή ενισχύουμε το μηχανισμό MPCC, ε, θα ήταν χρήσιμο να ενισχύσουμε και τη δυνατότητα σχεδιασμού και συντονισμού μεταξύ της ιεραρχίας της στρατιωτικής και πολιτικής κάθε φορά. Έρχομαι τώρα στο σχέδιο εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Παγκόσμιας Στρατηγικής. Πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πολλή δουλειά και από σας και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια ε, νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνα στην Ευρώπη. Το Δεκέμβριο του 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, ενέκνε μια αυξημένη φιλοδοξία για την άμυνα και την ασφάλεια, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να διαδραματίζει το ρόλο της ως αξιόπιστος ε, πάροχος ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την εφαρμογή και εκτέλεση της παγκόσμιας στρατηγικής, έχει προβληθεί πάρα πολύ αλλά εξαρτάται από τη δυνατότητα και τις ικανότητε που διαθέτουν τα κράτη-μέλη. Πολύ σύντομα τώρα θέλω να αφαιρθώ ε, σε μερικά από τα εργαλεία που έχει αυτή η στρατηγική. Πρώτο, η πολύ γνωστή μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, ΠΕΣΚΟ, η οποία έχει στόχο να διευρυνθεί, να εμβαθυνθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και να είναι πιο ολοκληρωμένη. Είναι ένα από τα εργαλεία. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ε, δημιουργία ικανοτήτων, αλλά και τη δέσμευση για τις αποστολές και τις επιχειρήσεις και έχει άμεση επίπτωση ε, στις αποστολές και τις επιχειρήσεις. Ε, το επόμενο διάστημα πέρα από τα πολλά συνεργατικά προγράμματα, 30 το σύνολο, έχουμε 25 κράτη-μέλη από τα 28 που έχουν δεσμευθεί. Η μετάβαση ε, από το στάδιο της ίδρυσης της ΠΕΣΚΟ μέχρι να δώσει αποτελέσματα θα είναι αυτή που θα, δώσει, θα δείξει την πραγματική αξία. Έχουμε μια καλή ευκαιρία τώρα για να μετρήσουμε ε, τον αντίκτυπο ένα χρόνο μετά την εφαρμογή της ΠΕΣΚΟ. Άλλο ε, εργαλείο η συντονισμένη ετήσια αναθεώρηση της άμυνας, CARD, για να ε, συγχρονίζεται καλύτερα και να προγραμματίζεται καλύτερα η στρατιωτική δραστηριότητα. Αυτό θα διευκολύνει το συντονισμό των δυνάμεων, των προσπαθειών και ε, τα κοινά ε, έργα και προγράμματα. Το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αμυντικής Έρευνας δίνει χρηματοδότηση σε επιλέξιμα σχέδια για την άμυνα. Αναφέρθηκα λίγο στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για την Ειρήνη, που είναι σημαντική πρωτοβουλία με στόχο να ενισχύσει τη δυνατότητα ασφάλειας και άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διευκολύνει την επόμενη γενιά. Ένας μηχανισμός χρηματοδότησης ε, ενώνει τα διάφορα μέσα χρηματοδότησης που είχαμε μέχρι τώρα για να αξιοποιούνται καλύτερα και να διευρυνθεί και το πεδίο εφαρμογής τους. Έχει συνεισφέρει πολύ στην ανάπτυξη των απαραίτητων στρατιωτικών ικανοτήτων για να φτάσουμε στο συμπεφωνημένο επίπεδο ε, φιλοδοξιών. Είναι πολύ σημαντικό να ε, ανταποκριθούμε στα ε, όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Ε, υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από μη ε, Ευρωπαίους εταίρους να συμμετέχουν στην ΕΠΑ. Ε, στις αρχές του Νοεμβρίου 2018 που ανέλαβα, ε, ε, αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θεωρώ απαραίτητο να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις ε, στην έννοια της στρατηγικής αυτονομίας που απορρέει από την παγκόσμια στρατηγική. Σε ό,τι αφορά αυτό και την το πώς ε, συνδέεται με το πλαίσιο της ΕΠΑ. Ε, γνωρίζω ότι χρησιμοποιείται αυτή η έννοια σε πολλά διαφορετικά φόρα και μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες παρανοήσεις και άχρηστες συγκρούσεις γνωρίζουμε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ και με μια κοινή διακήρυξη του Ιουλίου 2016 αλλά και του Ιουλίου 2018. Στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μας για να προωθούμε την ασφάλεια ε, και την ειρήνη στον Ατλαντικό. Ωστόσο, παρά το γεγονό ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη τη Ένωση είναι μέλη του ΝΑΤΟ και καταβάλουν κοινέ προσπάθειε οι δύο οργανισμοί να εμβαθύνουν τη συνεργασία του, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη έχουν αρχίσει μια διαδικασία ε, καθορισμού δικών τους στρατηγικών στόχων. Και τώρα βλέπουμε τα επιτέγματα. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Ούτε στόχος είναι να ανταγωνιστούμε το ΝΑΤΟ. Ε, απλώς έχει νόημα γιατί οι δύο οργανισμοί έχουν κοινέ αξίε, κοινά ε, συμφέροντα και κοινά μέλη εμπολής. Αλλά θα πρέπει λοιπόν να είναι συμπληρωματική η δράση μα με την Ατλαντική Συμμαχία. Ε, δεν ε, είναι Ε, τώρα ε, αυτό ένα παιχνίδι όπου όταν αυξήσουμε τις ικανότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι θα πάρουμε από το ΝΑΤΟ και θα αφαιρέσουμε κάποια στοιχεία. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας. Είναι βασικός στρατηγικός στόχος του ίδιου του ΝΑΤΟ. Και το ζητούν και οι ίδιες οι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι σαφές ότι η αμυντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπονομεύσει το ΝΑΤΟ, μόνο να το ενισχύσει. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι στρατιωτικές ικανότητες είναι κτήμα ε, των ευρωπαϊκών κρατών μελών και των συμμάχων τους. Η στρατηγική αυτονομία λοιπόν δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτονομία ή ανεξαρτησία από κάτι ή από κάποιον άλλον, δηλαδή όπως είναι το ΝΑΤΟ, αλλά αυτονομία για δράση, για να δρούμε ε, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις από την παγκόσμια στρατηγική μας. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να έχει μεγαλύτερη αυτόνομη ικανότητα να εκτελεί ε, ευρύτερης κλίμακας στρατιωτικές αποστολές με τους εταίρους όπου και όποτε ε, είναι δυνατό αλλά και όταν είναι απαραίτητο. Υπάρχει μια εργαλειοθήκη της ΕΠΑ ε, που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καλύτερη, περισσότερη επιρροή και παρουσία και στις αφρικανικές χώρες αλλά και με άλλους εταίρους ή άλλε οργανώσεις όπως είναι το ΝΑΤΟ. Παράδειγμα, στρατιωτική κινητικότητα, οι μεταφορές. Ε, εξαιρετική συνεργασία έχουμε ε, και συμπληρωματική ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Ήδη στα πρώιμα στάδια για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων ε, ό,τι αφορά τις υποδομές, τα οχήματα και τα λοιπά. Έχουμε μόνιμη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και πάγια και αυτό φαίνεται ε, και από τις σχέσεις που έχουν οι δύο στρατιωτικές επιτροπές. Υπάρχει αμοιβαία και μόνιμη ανταλλαγή ε, ενημέρωσης με ε, εστίαση στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι υψηλή προτεραιότητα και για τους δύο οργανισμούς. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνω λέγοντας δύο λόγια για την ε, Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ. Συμμετέχουμε άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα. Ε, βασικό στόχο έχουμε να συμβουλεύουμε το πολιτικό επίπεδο, ε, διαβιβάζοντας τις απόψεις των αρχηγών γενικών επιτελείων. Η παγκόσμια στρατηγική περιγράφει ε, το όραμα μιας ισχυρότερης Ευρώπης και περιγράφει και τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιόπιστη, υπεύθυνη και δυναμική. Δεν μπορούμε βέβαια μια ανοιχτή να ε, οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη, ούτε με ε, ούτε χωρίς να επενδύουμε στους απαραίτητους πόρους, που είναι χρόνος, χρήμα, πολιτικό κεφάλαιο και ανθρώπινο κεφάλαιο. Χρειάζεται υπομονή και μακροχρόνιος σχεδιασμός. Η στρατηγική αυτή μας έχει δώσει ένα ε, σχέδιο. Τώρα εναπόκειται στα κράτη-μέλη, αν θέλουν να συνεχίσουν σε αυτή τη γραμμή, να είναι πιο αποτελεσματικά, να ανταποκριθούν καλύτερα, χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα και διαθέσιμα εργαλεία, ή εάν ε, προτιμούν να ε, επιστρέψουν σε ένα πιο παθητικό ρόλο για να ε, αποφασίσει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, για τα οικονομικά. Εγώ δεν υποτιμώ την οικονομία, αλλά έχει δείξει ότι είναι περιορισμένη η δυνατότητα της να επηρεάσει τα παγκόσμια ε, τεκτενόμενα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο διπλωματία και ανθρωπιστική βοήθεια. Με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ολοκληρώνονται όλα αυτά τα μέσα που έχει με στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές και επιχειρήσεις επιτόπου γνωρίζετε ότι η στρατιωτική πτυχή είναι αναπόσπαστο τμήμα της ασφάλειας και της άμυνας κάθε κράτους μέλους. Φιλοδοξία μας λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να χρησιμοποιούμε τις στρατιωτικές ικανότητες με πιο ακριβή τρόπο και πιο συνεκτικό για να εφαρμόσουμε την παγκόσμια στρατηγική. Για να το επιτύχουμε αυτό χρειαζόμαστε τα εξή τρία και έχουμε αρχίσει να τα χτίζουμε. Μια ισχυρή ιεραρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, διαλειτουργικές ένοπλες δυνάμεις και ισχυρά οικονομικά μέσα. Θα πρέπει να συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας εκεί, χωρίς να χαλαρώνουμε, ε, προσιλωμένοι στην Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική και στην ισχυρότερη Ευρώπη. Τούτων όλων λεχθέντων, ελπίζω να σας διαφώτισα ε, και να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ε, σα δίνω και πάλι το λόγο για οποιασδήποτε για αυτή την παρουσίαση, στρατηγέ. Και τώρα αρχίζει η ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές. Δύο ερωτήσεις καταρχήν από, μέρου μου. Η εντολή αυτή τη στιγμή της αποστολής Σοφία θα εκπνεύσει πολύ γρήγορα. Τι βήματα θα πρέπει να αναλυθούν ούτως ώστε να τονώσουμε την ασφάλεια περαιτέρω στη Μεσόγειο. Και ποια είναι η συμβουλή σας προς την ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τη σύγκρουση. που υπάρχει στη θάλασσα του Αζόφ. Ο κύριος Γκάλερ θα πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πολύ πλήρης παρουσίαση, πολλά θέματα θέσατε, πολλές ερωτήσεις ε, για την Άλθια. Είναι η μόνη αποστολή όπου ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναλάβει από κοινού δράση. Ξεκίνησε πάρα πολύ παλιά. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια προβλήματα, κάποιες ε, αναταραχές εντός της Βοσνίας και Ζεγοβίνης. Ε, επειδή έχουμε στρατεύματα επιπλέον, αλλά και έχουμε και κάποιες μονάδες stand-by εκτός της Βοσνίας ε, Ζεγοβίνης. Έχετε κάνει κατάρτιση και εκπαίδευση για να μπορούμε να μεταφέρουμε αυτές τις δυνάμεις. Και επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ε, Βοσνία, δεν θα πρέπει αυτά τα στρατεύματα που είναι εκτός να μπουν στη Βοσνία. Για τη Σοφία τώρα, αυτά τα προηγούμενα ήταν για την Αλθεία. Η διοίκηση ε, βρίσκεται στην Ιταλία αν δεν απατώμε. Έχουν στείλει... Οι Γερμανοί μάλλον αποσύρθηκαν από εκεί. Ε, άρα έχουν μείνει μόνο τους Ιταλοί με τους, ε, με, τους πρόσφυγες. Ε θα προσπαθήσουν να τους προωθήσουν στην ε, Λιβύη. Αλλά οι Λίβοι δεν κάνουν τίποτα, ας πούμε. Ενδεχομένως και ο κ. Σαλβίνη θέλει να υπάρξουν κάποια, θέλει να υπάρξουν κάποια θύματα, ούτω ώστε να υπάρξει αποτρεπτικό, το αποτρεπτικό στοιχείο για τους υπόλοιπου που θα διανοηθούν να περάσουν τη Μεσόγειο. Πάντω το θέμα ε, δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει, παρότι η αποστολή ίδια έχει τελειώσει. Για τον Northwood είπατε ότι υπάρχει θέμα με μετεγκατάστασης ε, στην Ισπανία από το Ηνωμένο Βασίλειο και μέρη στη Βρέσδη. Οι Βρετανοί έχουν προσφέρει οτιδήποτε ως μη μέλη, ας πούμε, έχουν πει ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν ε, παρόλα αυτά. Και εμείς έχουμε προσφέρει κάτι στους Βρετανούς. Σε περίπτωση που υπάρξουν κάποιες ε, αποστολές, ας πούμε, follow-up, ε, στις οποίες θα μπορούσε να βοηθήσουν. Στις αποστολές κατάρτισης. Είπατε ότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμωρήσουμε τα κράτη-μέλη τα οποία πολιτικά έχουν συμφωνήσει με αυτές τις αποστολές αλλά δίνουν τις απαραίτητες δυνάμεις. Έχετε απάντηση για αυτό το θέμα. Ή εμείς πρέπει να στυλιτεύσουμε κάποια κράτη-μέλη, ας πούμε. Ο μηχανισμός για τη διευκόλυνση της ειρήνης ε, που προβλέπετε. Κάποια κόστη θα μπορούσαν να χρηματοδοθούν μέσω αυτού του μηχανισμού. Ο μηχανισμός Αθήνα εντάχθηκε σε αυτόν τον ειρηνευτικό μηχανισμό και υπάρχει περίπτωση για κοινό προϋπολογισμό. Εγώ θα έλεγα να επιμεριστούν τα κόστη, ούτως ώστε να είναι πρόθυμα και περισσότερα κρατημέλη να βοηθήσουν. Είναι σωστός τρόπος ε, αυτός λοιπόν. Πρέπει να αντικαταστήσουμε την ε, Αθηνά με, την ε, Ευρωπαϊκή, με τον Ευρωπαϊκό Αυτομηχανισμό για τη διατήρηση της ειρήνης. Ο κύριος Πάσκου, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Μιλάμε για μια τεράστια παλέτα ας πούμε, συμφερόντων και θεμάτων που μας απασχολούν και τα οποία θίξατε. Δύο ερωτήσεις από πλευράς μου. Οι Αμερικανοί καταρχήν πάντα μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνά μας. Και όταν το κάνουμε αυτό, αρχίζουν να έχουν υποψίες. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Κάθε φορά λοιπόν πρέπει να δίνουμε εξηγήσει. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσουμε οτιδήποτε. Έχουμε έναν διάλογο στρατιωτικό, α πούμε, με του στρατιωτικού Αμερικανού ομόλογους σα, ούτω ώστε να του δείχνετε έμπρακτα ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να έχουν υποψίε απέναντί μα Και δεύτερον, Πόσο παρακολουθείτε την κατάσταση ε, και στη θάλασσα του Αζόφ, αλλά και γενικότερα στην Μαύρη Θάλασσα. Μια ναι, και είναι χώρος που ανήκει στην, στις αρμοδιότητες του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στους πανελίστες. Εκτός αν υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις. Σας βλέπω λοιπόν. Σας δίνω το λόγο. Ο κύριος Ντρογεύσκη. Ευχαριστώ. Ο στρατηγός ε, ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και κάποιες προσπάθειες που κάνουν τα κράτη-μέλη ε, και μας περιγράψατε την κατάσταση από τη σκοπιά της Στρατιωτικής Επιτροπής. Αλλά μιλήσατε και για μια νέα προσέγγιση ε, στα μελλοντικά σχέδια. Και θα σας παρακαλούσα, στρατηγέ, πάρα πολύ σύντομα να μας ε, πείτε ε, τι αλλαγές να περιμένουμε. Τι αλλαγές έχετε υπόψη εσείς στη Στρατιωτική Επιτροπή. Ευχαριστώ. General, sir, I think that's the end. Ευχαριστώ. Τέλειωσαν εδώ οι ερωτήσεις. Τώρα ο στρατηγός θα απαντήσει και θα κάνει άλλες παρατηρήσεις εφόσον το επιθυμεί. Thank you. Thank you. I start with... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω με τη Σοφία, λοιπόν. Ξέρετε πως η εντολή κλείνει 31 Μαρτίου. Λίγη. Και πρέπει να σας πω πως πήγα στο Βουκουρέστι πρόσφατα και εκεί όλοι οι Υπουργοί Άμυνας μου επανέλαβαν πόσο σημαντική είναι αυτή η αποστολή, την εντολή της αποστολής που είναι να ε, παρεμποδίσει αυτά τα ε, δίκτυα ελαθρομεταναστών, ε, να επιβάλλει το εμπάργκο όπλων στις λιβικές ακτές. Οπότε καταλαβαίνετε πως υπάρχουν και κάποιες δευτερεύουσες επιπτώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις δράσεις εκεί και σύμφωνα με τα όσα λέμε εμείς οι στρατιωτικοί θα πρέπει η επιχείρηση Σοφία να συνεχίσει. Είναι πολύ σημαντική για την οικοδόμηση δυναμικού επίσης. Είναι κάτι πολύ συνεκτικό με την σφαιρική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια υποδειγματική ε, επιχείρηση που μπορεί να ενισχύσει τη θέση μας και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και τα επόμενα στάδια γιατί χρειάζεται η συνέχεια για να περάσουμε στη δεύτερη φάση να εγκριθεί από τον ΟΗΕ Δεν μπορώ βέβαια εγώ να προδικάσω ποια θα είναι η πολιτική απόφαση. Πάντως πιστεύω θα ήταν ε, ένα πραγματικά αμφιλεγόμενο και μη ορθό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένων των προσδοκιών των χωρών της Αφρικής αν λέγαμε πως είναι αδύνατο να βρεθεί μια λύση για να συνεχιστεί η αποστολή αυτή, γιατί θα δίναμε την εντύπωση της διέρεσης, κάτι το οποίο θα είχε μάλλον αρνητικές επιπτώσεις για τη σφαιρική ε, στρατηγική και για την εταιρική σχέση με τις άλλες όχθες Μεσογείου. Γιατί ξέρετε πως η κεντρική Μεσόγειος αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα και θα παραμείνει πρόβλημα γιατί θα είναι η βασική οδός για τους μεταναστενές. Και στην Άκαμπα μου το είπε κάποιος πρόσφατα και το ξέρω γιατί 10 χρόνια ασχολούμαι πως το πρόβλημα των μεταναστών έχει αυξομοιώσεις μεν, αλλά είναι εκατομμύρια που επηρεάζονται, οπότε η Ευρώπη πρέπει να βρει μια λύση με αλληλεγγύη Δεν ξέρω και τι θα γίνει. Για τα τεχνικά εμείς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε. Στο πολιτικό επίπεδο αυτό δεν μας ε, αφορά. Για την θάλασσα του Αζόφ και τη σύραξη εκεί δεν είναι αυτή τη στιγμή ε, το λιμάνι ε, στρατιωτικό θέμα. Το παρακολουθούν οι πρέσβεις εκεί. Γίνονται και κάποιες συναντήσεις ενημέρωσης με πληροφορίες για να γνωρίζουμε πώς έχει κατάσταση. Παραμένουμε λοιπόν στη δήλωση του πολιτικού επίπεδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βρεθεί μια λύση. Και είναι πολύ σημαντική η σχέση μας γιατί στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης με τις ανατολικές χώρες θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την αμοιβαιότητα και την εμπιστοσύνη με τις χώρες αυτές. Εδώ πρέπει να σας πω πάντως πως ε, μάλλον το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάσταση πιο πολύ. Αλθέα είναι η μοναδική μεικτή επιχείρηση με το ΝΑΤΟ και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική. Πιστεύω πως είναι καθήκον μας να αυξηθεί η συνέργεια και οι, κοινέ δράσεις με τον ΝΑΤΟ και με τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, ε, για τις σχέσεις με τον ΝΑΤΟ, συμφωνώ και εγώ, θα πρέπει ε, να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ ε, τη βοήθειά σας και είναι μια εκτελεστική αποστολή και έχουμε αποφασίσει να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο γιατί έχει τη δυνατότητα να διευρύνει πεδίο και στόχους σύμφωνα με τις εξελίξεις στο πεδίο κυρίως για, τους, ε, για τις εφεδρίες που είναι σημαντικές και ξέρω πως πέρσι οι εφεδρίες, το τάγμα εφεδριών ανέλαβε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη να σας πω πως μας είχαν πει εκεί δυνάμεις πως ε, έχουμε καθήκον συμμετοχής για να συνεχίσουμε με τα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει εκεί. Ah, eh, about Και για το Ηνωμένο Βασίλειο να σας πω πως πολύ ενδιαφέρονται και τα όσα ακούστηκαν. Θα δούμε. Θα συνεχίσουν οι συζητήσεις στα πλαίσια του Brexit. Νομίζω 12 το μεσημέρι, 31 Μαρτίου, κλείνουν. Άρα λοιπόν για να γίνει μετέρη θα χρειαστεί ένα πλαίσιο συμμετοχής, μια συμφωνία για να έχουμε το δικαίωμα να ανταλλάσσουμε απόρριτες πληροφορίες. Καταλαβαίνετε πως αυτό πρέπει να συζητηθεί μετά τις πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει και σε άλλες αποστολές, Αλθέα για παράδειγμα και εκεί η συμμετοχή των Βρετανών και προσφέρουν ε, δυναμικό και από τη στιγμή που θα φύγουν θα πρέπει να υπάρχει το συντομότερο δυνατόν συμφωνία για να έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν να συμμετέχουν όπως σίγουρα επιθυμούν. Τώρα, για τις ΕΠΑ έχουμε άμεσες επαφές. Καμιά φορά είναι πιο εύκολο να συζητήσει κανείς το τι συμβαίνει στο δικό μας επίπεδο και κατανοούν πως σε επίπεδο αποστολών μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανα μια συνάντηση στην οποία συζητήσαμε τη Σομαλία και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πολύ σημαντικός και μοναδικός εκεί όπως επίσης στην περιοχή του Σαχέλ της Αφρικής και να σας πω πως αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο εύκολο να βασιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στο ΝΑΤΟ. Εγώ ήμουν αξιωματικό και είμαι πολύ, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό στο ΝΑΤΟ πολλά χρόνια, αλλά από το 2011 και μετά πρέπει να σας πω πως το ΝΑΤΟ ασχολείται με τη συλλογική άμυνα και εμείς θα πρέπει να είμαστε συμπληρωματικοί ως προς αυτή του τη δράση. Πιστεύω προσωπικά και βέβαια εγώ δεν μπορώ τώρα να ε, αναφερθώ σε πολιτικές ε, υποθέσεις που μπορεί να γίνονται, αλλά πρέπει να σας πω πως πιστεύω πως χρειαζόμαστε μεγαλύτερη στήριξη από τους ε, στρατιωτικούς κύκλους. Εγώ ζητώ παραπάνω χρήματα και ελπίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα προσφέρει έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο εξοπλισμό, περισσότερη διαλειτουργικότητα, καλύτερο δυναμικό, περισσότερες ε, δυνατότητες να αποκριθούμε σύμφωνα με το δυναμικό το οποίο έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Εκπαιδευτικές αποστολές. Τρεις γίνονται αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία εκτελεστική επιχείρηση σε κάποιες από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου. Μογκαντήσου, Μαλή, ε, Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ελπίζω πως θα συνεχίσουν να κάνουν αυτή την εξαιρετική δουλειά. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τους δώσουμε καλύτερες συνθήκες για να συνεχίσουν. Ε, στο Μαλί, για παράδειγμα, 500 άτομα, 550 ε, περίπου, Εκεί η δική μας είναι γύρω στους 50 στην ποσόστοση. Πολλά πρέπει να κάνουν. Συντονισμό, συνεργασία και όταν ήμουν ε, επικεφαλής στην ε, UNIFIL στο Λίβανο. Είχα ε, γύρω στα χίλια άτομα πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που έπρεπε να συντονίσω και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως χρειάζεται μια ισχυρή εντολή έτσι ώστε αυτός ο συντονισμός να γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης, μηχανισμός για την ε, ειρήνευση. Για να είναι πιο αξιόπιστες αυτές οι αποστολές. Γιατί εμείς ε, εκπαιδεύουμε τους Σομαλούς. Βέβαια, αυτή η εκπαίδευση γίνεται χωρίς να έχουν ούτε επαρκή βενζίνη για την εκπαίδευση, ούτε υπαρκή ε, ε, πυρομαχικά και αυτά μπορούν να αποκτηθούν μόνο σε διμερές επίπεδο, όχι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αν μπορούμε να αναλάβουμε από κοινού το κόστος, τότε η δική μας εκπαίδευση θα είναι πιο αξιόπιστη, κάποια άλλα μη ε, ευρωπαϊκά κράτη μπορεί να μην μας αγκαλιάσουν αλλά στην αρχή είχαμε τρίτε χώρες που θα ήθελαν πάρα πολύ να συνεργαστούν μαζί μας, αλλά επειδή δεν έχουν τη χρηματοδότηση, δεν είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής. Οπότε αν ανοίξουμε αυτή τη ε, ε, δυνατότητα θα καταλήξουμε σε μια υποφελή για όλους συνεργασία. Δηλαδή ε, κάτι που να συνδυάζει την επιχείρηση Αθήνα, όπως επίσης και το μηχανισμό για τη χρηματοδότηση ε, για την Αφρική. Εγώ ήμουν και στο πεδίο διοικητής για πέντε χρόνια και πιστεύω ότι αν κάποιος δείξει αξιοπιστία όλοι τον ακολουθούν. Αν απλώς δίνουμε οδηγίες ε, χωρίς κάτι παραπάνω, οι προσπάθειές μας θα μείνουν ημιτελείς. Καμιά φορά αυτό είναι ε, εκνευριστικό, αλλά ξέρετε, έχω αναλάβει εδώ την Προεδρία εδώ και τρει ε, μήνε. Έχω μεγάλο θαυμασμό για το τι έγινε μέχρι σήμερα. Καμιά φορά για μένα είναι και λίγο δύσκολο να κατανοήσω πώ είναι δυνατόν να έχουμε προβλήματα στη δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, να βρούμε ε, ε, κονδύλια για το μικρό στρατιωτικό νοσοκομείο που χρειαζόμαστε για την αποστολή. Πρέπει λοιπόν και εγώ να τα πάω καλύτερα στο στρατιωτικό περιβάλλον που υπάρχει. Γιατί ξέρετε πως υπάρχουν πολλά στοιχεία που τρέχουν. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει ε, η αποστολή αυτή να ε, είναι πετυχημένη, να φανεί η Ευρώπη πετυχημένη. Και επειδή τώρα μιλάμε για λίγοι, δύο, τρεις δεκάδες ανθρώπους, είχαμε μία περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μας είχαν τη δυνατότητα να στείλουν χιλιάδες, χιλιάδες άτομα. Και επιστρέφω στα παραδείγματα του 2006, όταν δημιουργήθηκε η UNIF, μέσα σε 15 μέρες τα ευρωπαϊκά κράτη στα πλαίσια της αποστολής αυτής του ΟΗΕ αποφασίστηκαν στα, στη συνάντηση που έγινε υπό τον Κόφι να στείλουν 6.000 προσωπικό μέσα σε μέρες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό για να καταλάβουμε ε, τη σημασία που έχει για την Ευρώπη και αυτή τη στιγμή νομίζω δεν υπάρχει και αναλλακτική λύση για μας. για την ε, Μαύρη Θάλασσα. Αυτά που είπα και προηγουμένως και θα ήθελα να σας ακούσω ξανά γιατί πρέπει να σας πω ότι βάζοντας τα ακουστικά έχασα το πρώτο κομμάτι οπότε μάλλον δεν άκουσα ολόκληρη την ερώτησή σας. Ο κύριος Δρογεύσκη παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έλεγα λοιπόν ε, ότι ε, αναγγείλατε κάποιες αλλαγές στο μέλλον. Τι αλλαγές είναι αυτές. Ναι, τι αλλαγές θα κάνετε στο μέλλον. Α. Για το μέλλον είμαι αισιόδοξο. Ε, ε, Ξέρω ότι η διεθνής κοινότητα έχει αποκτήσει εμπειρία Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλέ προσδοκίε από την Ευρώπη ε, στη Σομαλία και σε άλλε τρίτε χώρε. Το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κινητοποιήσει πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά στοιχεία, ότι έχει την αξιοπιστία, μπορεί να κάνει πολιτικές αποστολές ε, με την υποστήριξη κάποιων στρατιωτικών επιχειρήσεων, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στρατιωτική οργάνωση, έτσι. Αυτό γεννά πάντως πάρα πολλές προσδοκίες. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλύει και μπορεί να επιλύσει πολλά ευρωπαϊκά προβλήματα και αυτή τη στιγμή που είχαμε τόσες αλλαγές και που αναδιαρθρώνονται πάρα πολλές οργανώσεις, ακόμα και το ΝΑΤΟ ανα διαρθρώνει ας πούμε, την κοινή δομή και ξαναβλέπει την, το δόγμα της συλλογικής άμυνας, είναι πολύ σημαντικά αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ στο ΝΑΤΟ ήμουν το 2011. Ήμουν στη συνάντηση της Λισαβόνας, όταν το ΝΑΤΟ άλλαξε και συρρυκνώθηκε. Πριν λίγα χρόνια επίσης ε, αντέστρεψαν αυτή την αλλαγή που είχαν αποφασίσει το 2011, την ακύρωσαν. Κατά πάση πιθανότητα, οι νατοικές δυνάμεις θα ξαναδράσουν στο εξωτερικό σε περίπτωση κρίσης, ε, για διαχείριση των κρίσεων. Το μέλλον είναι στην ε, οικοδόμηση του δυναμικού. Να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία όπου υπάρχει αστάθεια, τις περιοχές αστάθειας, για να είμαστε σε δράση να επιχειρήσουμε. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, παγκόσμια στρατηγική της, με τον Global Strategy, μπορεί να δώσει μια απάντηση. Το βασικό είναι να υπάρχει η συνένεση από τα 28 κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ο στρατηγός πρέπει να φύγει στις 12 ακριβώς. Δεν χρειάζεται επομένω να κάνουμε νέο γύρο ερωτήσεων. Εάν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στο στρατηγό, να το στείλετε γραπτό. Αλλιώ τον ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Και έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος αυτής της νομοθετικής θητείας. Είμαι πεπισμένη ότι και, στο επόμενο, και με το επόμενο κοινοβούλιο θα Έχουμε πολύ συχνές ανταλλαγές απόψεων με τον επικεφαλής της ε, Στρατιωτικής Επιτροπής. Πάντα με χαρά σας βλέπουμε. Σας ευχαριστώ για την ε, πλήρη παρουσίασή σας και τις ε, ειλικρινείς απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Παρακαλώ να χειροκροτήσουμε τον στρατηγό. We start at... Σταματάμε και ξαναρχίζουμε στις 2.30 την απογευματινή μας συνεδρία.